Συνεχίζουμε την ε, συνεδρίασή μας, τα δε πρακτικά της 11ης Τρίτου και τα σχετικά κείμενα υπάρχουν διαθέσιμα, αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή ενστάσεις, επομένως αφού δεν υπάρχουν θεωρούμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Και τώρα